τα οποία μπορούμε να έχουμε από τις απορρίψεις έτσι ώστε να καλύψουμε και επιπλέον ανάγκες αυτού του προγράμματος. Ευχαριστώ Επίτροπε. Εφόσον ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις έχουν κατατεθεί τέσσερις αιτήσει ε, ψηφισμάτων που θα ψηφιστούν ε, σήμερα στις 12 και έκλεισε η συζήτηση από αυτού του σημείου. Τώρα έχουμε ε, την έκθεση DAF σχετικά με την τροποποίηση της πράξης επί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταρχήν το λόγο έχει ο κύριος DAF για 5 λεπτά. Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συνοψίσω ε, τα βασικά στοιχεία του μεταρρυθμιστικού πακέτου το οποίο συμφωνήθηκε με μεγάλη δυσκολία σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε αυτή την ε, ε, ψηφοφορία διότι θα θέλαμε να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος με το Συμβούλιο σχετικά με την επανακατανομή των εδρών βάσει ενός μαθηματικού τύπου, ελπίζω, επί το οποίο φυσικά θα χρειαστεί να συμφωνήσουμε. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις ώστε να διευκολύνει την συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές αναμετρήσεις σε ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Η βασική πρόταση η οποία ήταν και σε κάποιο βαθμό αμφιλεγόμενη φυσικά, ήταν να έχουμε 25 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, βάσει μιας πανευρωπαϊκής εκλογικής ε, περιφέρειας ε, και διευρωπαϊκών ψηφοδελτίων καταλόγων μάλλον που θα καταρτίζονται από τα ευρωπαϊκά κόμματα. Ο στόχος είναι να τροποποιήσουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές αποδίδοντας κεντρικό ρόλο στα ευρωπαϊκά κόμματα για τις προεκλογικές εκστρατείες. Ε, εξατομικεύοντας, αν θέλετε, την ευρωπαϊκή διάσταση της προεκλογικής εκστρατείας. Ο διάδοχος ε, του Πρόεδρου Μπαρόσο ε, ίσως να εκλεγεί από μια διεθνική λίστα. Τα ευρωπαϊκά κόμματα θα πρέπει να ενηλικιωθούν επιτέλους. Τα περισσότερα εθνικά κόμματα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν πλέον να ε, υποστηρίξουν και να προαγάγουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με δημοκρατικό και αποτελεσματικό τρόπο. Μου λένε κάποιοι ότι δεν είναι ώρα τώρα για τέτοιες ε, ρίζοσπαστικές προτάσεις. Μα πότε είναι η κατάλληλη ώρα επιτέλους. στη, στον πολιτικό βίο ποτέ δεν είναι σωστή στιγμή. Για τίποτα. Η... Ε, αμφισβητείται τώρα η νομιμότητα του Κοινοβουλίου, οπότε εγώ κρίνω ότι είναι σωστή στιγμή να κινηθούμε. Τώρα θεσπίζουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Ε, λοιπόν, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ε, προωθήσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία, να την προβάλλουμε περισσότερο. Οι διαδηλωτές, οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα διαμαρτύρονται διότι υπάρχει αυτός ο δικοματισμός και έχουν... Ε, συγγνώμη, παραπονιούνται διότι ε, πρέπει να συμμετάσχουν και στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και κάποιοι ανησυχούν διότι θα αλλάξει το πρωτογενές δίκαιο για να υλοποιηθεί η πρόταση. Όμως η αλήθεια είναι ότι με ίσονο σημασία τροποποίηση της συνθήκης θα κάνουμε τις προβλέψεις για τους ε, Κροάτες βουλευτές ε, και θα ρυθμίσουμε την κατάσταση. Η παρούσα σύνθεση ούτως ή άλλως παραβιάζει την αρχή της συνθήκης ε, σχετικά με την αντίστροφη αναλογικότητα. Τη φθήνους αναλογικότητα. Μια άλλη καταγγελία που ακούμε, επιτρέψτε μου να στην εκθέσω, Ακούγονται επικρίσεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν ε, βουλευτές σε δύο τάξεων, δύο κατηγοριών. Ε, οι στάρ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι υποδέστεροι, ε, οι όσοι βουλευτές δηλαδή θα εκλέγονται βάσει των εθνικών καταλόγων. Πλην όμως η συνθήκη προβλέπει ότι είμαστε αιρετοί εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και θα πρέπει να παράσχουμε ε, τη δυνατότητα να γίνει η εκλογική μεταρρύθμιση αυτή, ώστε η συνθήκη ε, της Λισαβόνας ε, να μετουσιωθεί σε μια πολιτική δημοκρατική πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Ντάφ. Δέχεστε μια ερώτηση από τον κύριο Φόξ. Παρακαλώ κύριε Φόξ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ντάφ. Ο λόγος για τον οποίο η ψηφοφορία της εκθέσεώς σας έχει αναβληθεί είναι ότι η δική σας ομάδα, οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν ενιαία στάση στο εσωτερικό τους. Οι άλλες ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις. Δεν υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ μιας εθνικής εκλογικής περιφέρειας. Παρακαλώ γιατί δεν εγκαταλείπετε την πρότασή σας και να ψηφίσουμε ίσως κάποια πιο μετριοπαθή σημεία της εκθέσεώς σας να τα ψηφίσουμε. Κύριε Φόξ, εκτιμάτε με διαφορετικό τρόπο, αξιολογείτε με διαφορετικό τρόπο ε, τις απόψεις οι οποίες εκφράζονται στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων. Είναι αληθές ότι όταν κάποιος θίγει εκλογικού τύπου μεταρρυθμίσεις, τα μέλη αντιδρούν θεωρώντας ότι το θέμα είναι σχετικά θα έλεγα ευαίσθητο και μερικές φορές και σχετικά δυσάρεστο. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ακούσει προσεκτικά αυτά τα οποία εκφράζονται στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων να δούμε αν μπορούμε να τροποποιήσουμε την πρόταση, να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση και να της εμφυσίσουμε περισσότερο νόημα. Θα πρέπει όμως κύριε Φόξ να ξεκαθαρίσω ότι εγώ σαν εισηγητής θα εμείνω στην αρχή της Διεθνικής Εκλογικής Περιφέρειας. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει πάλι το λόγο η κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με ε, μία αναφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στο να μπορέσουν να, ένα μέρος των Ευρωπαίων βουλευτών να εκλέγονται από διεθνικές λίστες και αυτό δεν είναι ε, μία αναφορά στην έκθεση αλλά εις ε, την ε, αναφορά εις ε, την Ευρωπαϊκή Συνέλευση το 2002. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι οι πανευρωπαϊκές λίστες θα αναβαθμίσουν τις ευρωεκλογέ. Ας πω λοιπόν λίγα λόγια σχετικά με την έκθεση του κυρίου Άντριου Νταφ. Καταρχήν λαμβάνω υπόψη την προσπάθεια του εισηγητή και τον ευχαριστώ για αυτό ο οποίος επιζητεί ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο σε ένα τόσο δύσκολο θέμα. Η ουσία του εκθέσεως αναφέρεται ε, σε μια πανευρωπαϊκή λίστα όπου θα μπορούσαν να γίνουν οι εκλογές ε, στο σύνολο των 27 κρατών μελών. Είναι μια ιδέα την οποία αξίζει να επιζητήσουμε αλλά δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί και εδώ αρχίζουν οι ανησυχίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν λοιπόν δεν είμαι βέβαια ότι οι πολίτες θα καταλάβουν την ανάγκη να αυξήσουμε τον αριθμό των εδρών και αυτό ήταν το συμπέρασμα το, της ε, Ευρωπαϊκής Συνελεύσεως πάνω από τα 750 μέλη θα είναι δύσκολο να λειτουργήσει μία συνέλευση επίσης εάν αυξηθούν τα μέλη θα πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες εκτός και αν τα 25 επιπλέον ε, άτομα τα οποία ε, θα επιλεγούν στην ε, πανευρωπαϊκή λίστα έχουν ειδικό καθεστώς. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχετε ήδη διατυπώσει τροπολογίες για να αφήσετε την εναλλακτική αυτή λύση διαθέσιμη. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί κατανομής μεταξύ κρατών μελών και δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι σκόπιμο να ξεκινήσει τώρα, αλλά είναι βασικό θέμα εάν θέλουμε και τα 25 αυτά μέλη να αποτελέσουν μέλος του σώματος. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει κύρωση από όλα τα κράτη-μέλη και σε ορισμένα κράτη αυτό μπορεί να οδηγήσει έστω και σε δημοψήφισμα. Θέλουμε να διακινδυνεύσουμε μία αρνητική ψήφο τώρα, διότι υπάρχει μία κόποση με την Ευρώπη λόγω της οικονομικής λιτότητας και το δημοψήφισμα μπορεί να είναι επικίνδυνο και δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε μία αίσια έκβαση. Ε, έστω και μέσω το, της ψηφοφορίας στα κοινοβούλια. Γι' αυτό και προτείνουμε βάσει προτάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό είναι ένα σαφές ε, με ε, μήνυμα το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία δεν χρειάζεται να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι θα μπορέσει το Ευρωκοινοβούλιο να υποβάλει εγκαίρως μία πρόταση ε, για να εξεταστεί από το Συμβούλιο εγκαίρως πριν τις εκλογές του 2000. 12 κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε συγχρόνως να δημιουργήσουμε έναν ελεγκτικό μηχανισμό ο οποίος θα αποφεύγει τους διπλοψηφίσαντες διότι ίσως τα συστήματα αυτά θα είναι αναγκαία αφού κυρωθεί η αναθεωρημένη πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί χρόνο για να καταρτήσει την πρόταση της θα αργήσουν τα κρατη μελια να συμφωνήσουν, οπότε δεν βλέπω αυτό να μπορέσει να ολοκληρωθεί πριν από το 2019 και γι' αυτό ζητώ από την ε, Επιτροπή να παρουσιάσει μία αναθεωρημένη πρόταση για να ενθαρρύνει τους πολίτες να ψηφίζουν στις χώρες όπου διαμένουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνενεί αλλά η πρόταση αυτή έχει ε, μπλοκάρει στο Συμβούλιο από το 2006 διότι δεν υπάρχει ομοφωνία η οποία είναι απαραίτητη. Επίσης ένα άλλο θέμα αναφέρεται στις στατιστικές και στη ε, τη σύγκριση των στοιχείων σχετικά με τον πληθυσμό που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό επεξεργάζεται ένα σχέδιο προτάσεως η οποία σύντομα θα έρθει. Υπάρχουν και άλλα θέματα στην έκθεση αυτή και να είστε βέβαιοι ότι μπορούμε να δεχτούμε αρχές ε, όπως η καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών, ο σεβασμός των μειονοτήτων και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή συμφωνεί να γίνονται οι εκλογές το Μάιο αντί για τον Ιούνιο. Οπότε, κυρία Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι η έκθεση αυτή ε, επίση πραγματεύεται ε, ε, συνταγματικά θέματα πέραν των νομοθετικών και γι' αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη για τις εκλογές του 2014 για να προβεί σε ορισμένες αλλαγές στη διαδικασία. Προηγουμένως ανέφερα την την ε, τροποποίηση της ε, οδηγίας 93-109 για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε ε, τις υποψηφιότητες και να αποφύγουμε τις διπλές ψήφους όσον αφορά τις στατιστικές προετοιμάζουμε ήδη την πρόταση για να συγκρίνουμε καλύτερα τα στοιχεία σχετικά με τους πληθυσμούς και τέλος πριν τρεις μήνες ο Αντιπρόεδρος Έσκοβης σας πρότεινε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό νομικό καθεστώ για, τις ε, πολιτικές, για τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή εξετάζουμε τα θέματα κλειδιά στην έκθεση Γιαννάκου με ανοιχτό πνεύμα και ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σύντομα σας σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε που ε, χρειάστηκα τόσο χρόνο. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπη, σας ευχαριστώ που είστε τόσο ευαίσθητοι για το χρόνο που χρησιμοποιείτε και τώρα ακολουθούν οι ε, μιλητές εν των πολιτικών ομάδων και καταρχήν ο κύριος Σέπφιλιν για το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Ήταν ε, ξεκάθαρη η παρουσίαση τη ε, θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ όλου ιδιαίτερα τον Άντριο Ντάφ. Ήταν αγαστή η συνεργασία μα. Μία από τις προτάσεις της έκθεσης ε, για την άμεση εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιούργησε απρόσμενα μεγάλες προκλήσεις. Υπάρχει αντίσταση για, τον πανευρωπαϊκό, για την πανευρωπαϊκή λίστα που θα εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και θα ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ε, θα πρέπει να διερευνήσουμε την περαιτέρω το θέμα κυρίως επειδή είναι αμφιλεγόμενο και υπάρχει η πλειοψηφία που υποστηρίζει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ολκλήρωσης. Πώς γίνεται όμως ο πανευρωπαϊκός, η πανευρωπαϊκή λίστα τελικά να μην μπορεί να γίνει αποδεκτή ε, από πολλούς. Ε, εγώ θεωρώ ότι η αντίσταση αυτή πηγάζει κυρίως από αυτούς που είναι μάλλον κοντόφ οφθαλμοί και κοιτάζουν βραχυπρόθεσμα ε, τι συμβαίνει στην Ένωση. Αληθεύει αυτό. Δεν είναι, είναι αβέβαιο το μέλλον του ευρώ. Ζούμε αυτή την κρίση. Ακόμη προσπαθούμε να βρούμε μια λύση εξόδου από την κρίση. Όσοι εστιάζονται λοιπόν στα βραχυπρόθεσμα θα σας πούνε ε, δεν είναι ώρα τώρα να πειραματιστούμε ακόμη με το, την πανευρωπαϊκή λίστη, λίστα. Ε, ε, ε, η αντίθετη επιχειρηματολογία όμως είναι η ισχυρότερη. Ό,τι και να αποφασίσουμε απαιτείται περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όχι λιγότερη. Οπότε το ουσιαστικό θέμα είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την Δηλαδή η, καρδιά της δημοκρατίας είναι η εκπροσώπηση. Άρα αυτή η εκπροσώπηση θα πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της πανευρωπαϊκής λίστας, να εκπροσωπούνται οι πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο είναι κοντόφθαλμο και μάταιο να εστιάζουμε στα βραχυπρόθεσμα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε τώρα ε, από πλευρά ε, της ομαδα ε, ECR, ο κυριο Γκουαλτιέρη, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η σοσιαλιστική και δημοκρατική ομάδα θεωρεί ότι η οικοδόμηση ενός πραγματικού ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου είναι θα έλεγα βασική προϋπόθεση για να συνεχίσουμε στον δρόμο μιας πολιτικής Ευρώπης ικανής να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα και με κατάλληλα μέσα τις τεράστιες προκλήσεις τις οποίες μας δίδει αυτός ο αιώνας. Η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός ιδιαίτερα επί τη βάση των αρχών τις οποίες ανέφερε ήδη ο κύριος Νταφ που διευκρινίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες. Παρόλα αυτά και παρόλες όλες τις καινοτομίες της συνθήκης της Λισαβόνας και παρά την καθημερινότητα η οποία μας δείχνει πόσο απαραίτητη είναι η πολιτική Ευρώπη, η δημιουργία ενός ουσιαστικού πραγματικού ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου είναι κάτι το πολύ μακρινό. Η συζήτηση στα κράτη-μέλη είναι εσωστρεφής και εθνική. Τα πολιτικά κόμματα συζητούν, θα έλεγα, μονομερώς εθνικά τα προβλήματα και οι ίδιες οι ευρωεκλογές πάρα πολλές φορές παρουσιάζονται στους πολίτες σαν μία προέκταση της εσωτερικής πολιτικής συζήτησης και αυτό εξηγεί εν μέρη και την πολύ χαμηλή συμμετοχή. Εμείς θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Νόμου μπορεί να συνεισφέρει στον εξευρωπαϊσμό θα έλεγα τη συζήτηση γύρω από την πολιτική στην Ευρώπη. Δεν είναι βέβαια ο μοναδικός τρόπος για να το πετύχουμε αυτό. Έτσι λοιπόν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες γνωρίζοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται βέβαια Υποστηρίζουμε και την δημιουργία της Διεθνικής Εκλογικής Περιφέρειας. Υποστηρίξαμε όμως και την αναπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή γιατί απαιτείται να υπάρξει μεγαλύτερη ε, πλειοψηφία. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στην συνέχιση της προσπάθειας για την αλλαγή των εκλογικών ε, συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και τώρα για τους φιλελεύθερους η κυρία Τάιν ε, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, αγαπητέ Άντριου, καταρχήν εν ονόμα της πολιτικής μας ομάδας θέλω να σε ευχαριστήσω για την πολυετή εργασία την οποία έχεις αναλάβει και την ενέργεια με την οποία προσπαθείς να την επιβάλλεις γιατί κάποια μέρα Πρέπει να καταλήξουμε εκεί. Όπως το είπες και εσύ προηγουμένως, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Και πιστεύω ότι η χρονική στιγμή αυτή είναι κατάλληλη και θα πρέπει το Σεπτέμβριο να ψηφίσουμε την έκθεση διότι μετά θα χρειαστούν χρόνια ίσως δεκαετίες μέχρι ότου να μπορέσει να εφαρμοστεί αλλά πιστεύω ότι αν δεν ξεκινήσουμε τώρα δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε καν στην επόμενη δεκαετία. Εγώ προσωπικά προσωπικά θα ήθελα να το ζήσω επί των ημερών μου να βρεθώ σε ένα πραγματικό κοινοβούλιο με μια διευρωπαϊκή με ένα διευρωπαϊκό κατάλογο υποψηφίων γιατί αυτό είχαμε ζητήσει να είμαστε νομιμοποιημένοι όταν θα μας έχει ψηφίσει ε, ο κάθε ε, πολίτης Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή θα μπορεί να μας ψηφίσει. Ε, διαφορετικά θα μπορούσα να προτείνω μια συμβιβαστική λύση, δηλαδή για τα μικρά κράτη να μπορέσουμε να διευρύνουμε στο 10% τους υποψηφίους που θα συμπεριληφθούν στην πανευρωπαϊκή λίστα. Ε, Χθε συζητήθηκε αυτό και ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Δέχεστε μια μια ενδιάμεση ερώτηση από τον κύριο Στογιάννοφ. Κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Ένα κράτος το οποίο έχει ομοσπονδιακή δομή είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι φεντεραλιστές στην Ευρώπη ε, ονειρεύονται το αμερικανικό πρότυπο. Θέλετε να κάνετε μία ερώτηση, όχι μία ομιλία. Ναι, ναι, τώρα θα παρουσιάσω την ερώτησή μου. Στην κατάσταση αυτή λοιπόν δεν χρειαζόμαστε να είμαστε εδώ ιδιαίτερα φεντεραλιστές και δεν χρειάζεται να είμαστε πιο φεντεραλιστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να είμαι σαφής, ε, αυτή δεν είναι μία μέθοδος για να κάνετε μία ομιλία. Ε, εσείς ζητήσατε το λόγο, έχετε ζητήσει το λόγο και στο Catch the Eye. Θέλετε τώρα να διαγραφείτε από τη λίστα θα επανέλθετε, ε, διότι δεν ήταν ερώτηση και τώρα έχει τον λόγο ο κύριος Φόξ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κεντρική πρόταση της εκθέσεως ΔΑΦ είναι η δημιουργία 25 θέσεων ευρωβουλευτών που θα εκλέγονται από το σύνολο της Ευρώπης η δημιουργία μιας νέας εκλογικής ε, περιφέρειας για το σύνολο της Ένωσης ε, δημιουργεί προβλήματα σε επίπεδο δημοκρατίας. Σε ποιους θα είναι υπόλογοι αυτοί οι βουλευτές. Όχι βέβαια στους λαούς της Ευρώπης, θα είναι υπόλογοι μόνο στο Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα το οποίο τους τοποθέτησε στον κατάλογο αυτό. Θα μιλούν εξ ονόματος του κόμματός μου και του κόμματός τους και της ιεραρχίας του, όχι των λαών θα είναι μακριά από τους λαούς της Ευρώπης και θα αυξήσει την απόσταση ανάμεσα στον καθημερινό πολίτη και στην πολιτική στις Βρυξέλλες σήμερα. 25 επιπλέον βουλευτές θα κοστίζουν επίσης χρήματα και σε, επίσης ε, σε επίπεδο χρόνου και ε, γενικά ε, οικολογικό επίπεδο ε, χρειαζόμαστε 25 επιπλέον βουλευτές να ταξιδεύουν από τη μία άκρη στην άλλη αυτή της τεράστιας εκλογικής περιφέρειας. Θα δημιουργήσει προβλήματα και στους φορολογούμενους. Πώς θα ξοδεύουμε τόσα επιπλέον εκατομμύρια για επιπλέον πολιτικούς και το προσωπικό τους. Ο κύριος Νταφ θέλει επίσης μια νέα εκλογική αρχή για την εκλογή αυτών των επιπλέον βουλευτών. Όλες αυτές οι προτάσεις έχουν κοστολογηθεί φυσικά και όχι. Η τέλεση των εκλογών θα πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο των κρατών μελών. Πρόεδρε, οι μόνοι που ωφελούνται από, από τις προτάσεις αυτές είναι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ο κύριος Νταφ θέλει να δημιουργήσει αυτούς τους νέους βουλευτές μόνο και μόνο για να τους δώσει μία μικρή ανασχόληση. Η έκθεση Νταφ είναι μη δημοκρατική και έχει υψηλό κόστος, υπονομεύει την κυριαρχία των κρατών μελών και η πολιτική μου ομάδα είναι κατά. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. Τρεις μπλε κάρτες έχουν σηκωθεί. Θα δεχτείτε τις ερωτήσεις. 30 δευτερόλεπτα για τις ερωτήσεις σας, Σύγκλεα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε ε, Πρόεδρε. Ε, ναι μεν ε, αυτά τα οποία είπατε είναι σωστά αλλά συμφωνείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία στην οποία θα επευθυνόμαστε στις εκλογές και ένα γενικευμένο εκλογικό σύστημα. Είναι επικίνδυνο όμως αυτό και επειδή το κόμμα σας κυβερνά ή στην Αγγλία Αγγλία μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι θα μπλοκάρετε αυτό το θέμα. Την επόμενη ερώτηση έχει, ε, την επόμενη ομιλία θα κάνει ο κύριος Σμιτ. Κύριε Φόξ, νομίζω ότι και εγώ είμαι υπόλογο σε αυτούς οι οποίοι με ψήφισαν. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών που έχουν ψηφίσει ε, σε ένα κράτος ή στα 25 κράτη-μέλη. Δεν ε, είναι υπόλογοι, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, διότι εσείς σε ποιον αναφέρεστε. Και τελευταία ερώτηση του κυρίου Βίλαντ. Αγαπητέ συνάδελφε Φόξ, θα ήθελα να ξέρω πώς εσείς θεωρείτε ότι συμβιβάζετε ότι μόνο σε μελικά κράτη μπορούν να υποβληθούν υποψήφια από τα κράτη και οι ε, υποψήφια αυτοί είναι πιστοποιημένοι από την ε, κεφαλή του κόμματος στη χώρα σας παραδείγματος χάνει. Ο κύριος Φόξ έχει χρόνο να απαντήσει σύντομα. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω στην κυρία Σενκλέρ θα ήθελα να πω σαφώς ναι. Το Συντηρητικό Κόμμα θα μπλοκάρει την πρόταση αυτή. Στον κύριο Σμιτ θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι χρειάζεστε ένα σύστημα όπου θα μπορούσατε να διώξετε έναν βουλευτή που δεν σας αρέσει. Δηλαδή θα μπορούσα να τοποθετηθώ από το κόμμα μου αλλά θα μπορούσα να με διώξει η ψηφοφόρη μου πράγμα το οποίο δεν θα υπάρχει σε αυτό το σύστημα. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι για μένα κάθε κράτος, κάθε εθνικό κράτος πρέπει να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε όμως τώρα με τον ο κατάλογο των ομιλητών και τον λόγο έχει ο κύριος Χέφνερ για δυόμιση λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη χρειάζεται καινοτόμες ιδέες για να προχωρήσει. Ιδέες σύμφωνα με τις οποίες μια ευρωπαϊκή δημοκρατία θα μπορέσει να υλοποιήσει και θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια δημοκρατική Ευρώπη διότι λίγο επηρεάζουν οι πολίτες στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές συζητήσεις για ευρωπαϊκά θέματα και οι πολίτες πρέπει να έχουν επιλογή γιατί όπως είπατε αυτή είναι κυρίαρχη άρα χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό δικαίωμα πρωτοβουλίες χρειαζόμαστε μία αναθεώρηση του εκλογικού νόμου γιατί οι ευρωεκλογές είναι εθνικά θέματα μέχρι τώρα από εθνικά κόμματα με εθνικούς βουλευτές και ουσιαστικά για εθνικά διακυβέρνηση και πιστεύω ότι αυτό είναι παρανόηση των ευρωεκλογών διότι θα πρέπει να υπάρχουν άμεσες και έμεσες επιπτώσεις και με αυτόν τον τρόπο υποχρεώνει ε, κάποιος, θα πρέπει να μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να ε, υποβληθούν ευρωπαϊκά θέματα και ευρωπαϊκοί υποψήφοι. Επίσης θα μπορούσαν πλέον των εθνικών υποψηφίων να υπάρχουν και υποψήφοι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση διότι ποιον εκπροσωπούμε εδώ είμαστε απλώς μια ένωση των κρατών μελών και εκπροσωπούμε μόνο τα συμφέροντα των πολιτών της χώρας μας ή είμαστε εκπρόσωποι και μιας κοινή ευρωπαϊκής κοινότητας συμφερόντων και η αλήθεια είναι ότι είμαστε και τα δύο δεν πρέπει να παραβλέψουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο και αυτό ισχύει για τους πολίτες μας διότι υπάρχουν σε εκλογές και εθνικά θέματα αλλά και ευρωπαϊκά θέματα και προσβλέπω στην ημέρα όπου θα υπάρχουν δύο λίστες πέραν των εθνικών υποψηφίων με τους ευρωπαίους υποψηφίους και μέχρι στιγμής οι πράσινοι έχουν χαράξει νέο δρόμο διότι έχουν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έναν ευρωπαϊκό προεκλογικό αγώνα και αυτό το χρωστάμε στην Ευρώπη. Εάν θέλουμε λοιπόν κάποια μέρη να μπορέσουν οι Γερμανοί να ψηφίσουν Γάλλους υποψηφίους γιατί τους θεωρούν καλούς και το αντίστροφο πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ και τώρα για την Ηνωμένη η Αριστερά. Το λόγο έχει ο κύριος Ζόντεργαρτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τι η δημοκρατία? Το δικαίωμα του εκλεγήν μία φορά την πενταετία, όχι. Σε μία πραγματική δημοκρατία οι εκλογές είναι μία παρένθεση μέσα σε μία μακρά δημοκρατική διαδικασία. 25 επιπρόσθετοι βουλευτές θα ενισχύσουν τη δημοκρατία ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ε, θα μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στους ε, ψηφοφόρους ε, και τους ερετούς εκπροσώπους τους. Δεν νομίζω. Αυτή η πρόταση σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν αυξημένη εξουσία, θα έχουν περισσότερα ονόματα στα ψηφοδέλτια θα κατεβάσουν υποψηφίους που δεν θα προέρχονται από τη Μάλτα ή άλλες ε, μικρές χώρες. Ε, επικεφαλής ε, των ληστών θα είναι βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές από τη Γαλλία και από τη Γερμανία, από τις μεγάλες χώρες. Ευχαριστούμε κύριε Ντόφαλ. δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σας υποστηρίξω. Ευχαριστώ. Τώρα από πλευράς του EFD, e ο κύριος Αγνιού για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Έχω μία ερώτηση του κυρίου Λάινεν και πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το χρόνο. Ένα λεπτό σας παρακαλώ, με συγχωρείτε, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Εάν ε, θα πάρουμε αυτή την ερώτηση ακόμη και μετά πρέπει να συνεχίσουμε με τους ομιλητές και ε, μπορείτε να ζητήσετε το λόγο και να παρέμβετε στο Catch the Ο κύριος Λάινεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ο ε, καθένας να μία μπλε κάρτα και όχι ο ένας και ο άλλος καμία. Συμφωνώ ότι αν έχουμε ένα κατάλογο 25 υποψηφίων τότε αυτό ε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι από μία χώρα αλλά από 25 χώρες. Αυτό θα πρέπει να το καταρτήσουν τα πολιτικά κόμματα και εκεί θα υπερέχουν τα μικρά κράτη και όχι τα μεγάλα. Ο κύριος Ζόντεργκαρντ έχει το λόγο. Όχι, όχι, διαφωνώ κάθετα μαζί σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μια ευρωπαϊκή λίστα πώς ακριβώς ε, θα εκλεγούν αυτοί οι άνθρωποι, Πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν ε, στη Γερμανία σε σύγκριση παραδείγματος χάρη με τη Μάλτα ή στη, τη, τη Φινλανδία, ε, πόσοι υπάρχουν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την Κύπρο, είναι προφανές πως η πρόταση αυτή είναι ένα άλλο τέχνασμα ε, για να ενισχυθούν οι μεγάλες χώρες. Κύριε Άγνιο, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Τώρα έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι της έκθεσης είναι ε, το κομμάτι που αναφέρεται στη μείωση της προέως έλευσης σε ευρωπαϊκές εκλογές. Ε, πάνω από 60% ήταν παλιά και τώρα υπερβαίνει ε, το 40% κατά λίγο. Α, φοβερό επίτευγμα. Δείχνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τι πιστεύουν για το οικοδόμημά σας. Δεν τους αρέσει. Και εσείς τι απαντάτε. Αντί να αναρωτιέστε μήπως τους αρέσει καλύτερα η λιγότερη Ευρώπη, εσείς ναι, το ερμηνεύετε ως έτοιμα για περισσότερη Ευρώπη και θέλετε 25 επιπρόσθετους ε, βουλευτές που θα έχουν τις ε, υπερεθνικές ε, έδρες. Μα ποιος το θέλει αυτό. Στην Νότια Ευρώπη και στην Ιρλανδία βιώνουν όλοι την λιτότητα, φοβερές δυσχέρειες και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τόσο καταπληκτική η Ευρώπη. Τι γίνεται με την υπόλοιπη Ευρώπη θα ακολουθήσει καταστροφή γιατί αρχίζουν να έρχονται κύματα οικονομικών μεταναστών που πλήττουν και τις πλέον εύκολε χώρες ε, και έμεση επίπτωση είναι ότι τα κράτη-μέλη ε, ε, επανεγκαθιστούν τελωνιακούς ελέγχους στα σύνορα, κλειδονίζονται τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα εσείς αποφασίζετε ότι θέλετε περισσότερη Ευρώπη. Εγώ σταματάω και παρότι μου μένουν 15 δευτερόλεπτα γιατί θέλω λιγότερη Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τώρα. Ο κύριος Κόβατς από τους μη Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση του κυρίου Νταφ αναφέρεται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγνοώντας όμως ότι ε, οι πληθυσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδιαφορούν για αυτά τα όργανα. Εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μαθηματικούς τύπους για να λύσουμε το θέμα της εκπροσώπησης. Δεν γίνεται έτσι. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των νεοφιλελευθέρων, των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίες δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Και μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ήδη δυσκολεύεται η οργάνωση των εκλογών του 2014. και σύν της άλλης προτείνεται και μια νέα διεθνική εκλογική περιφέρεια, δημιουργώντας διαφορετικού τύπου πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορετικά επίπεδα εκπροσώπησης. Ο κόσμος αδιαφορεί και σε αυτόν τον κόσμο που αδιαφορεί του ζητάτε να ψηφίσει και εκλογικές περιφέρειες. Εσείς πιστεύετε ότι ένας Ούγγρος ψηφοφόρος ή ένας Γερμανός ψηφοφόρος ή ένας Βρετανός ψηφοφόρος, ένας θα ψηφίσει ένα Φιλανδό ή έναν Σουηδό, έναν βουλευτή τον οποίο δεν γνωρίζει. Κοιτάξτε, είμαστε 27 χώρες, 500 εκατομμύρια. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα με 25 βουλευτές να εκπροσωπήσετε όλους αυτούς. Νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει περισσότερη απόσταση από τις εκλογές. Ο επόμενος. Τώρα, επόμενος ε, το λόγο για δύο λεπτά, ο κύριος ε, Μέντες Ντεβίγκο. Ευχαριστώ. Ε, το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει τον εκλογικό νόμο και πρέπει να το πράξουμε διότι σύντομα θα υπάρχει μία νέα κατανομή εδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προσθήκη της Κροατίας. Γι' αυτό και συγχαίρω τον κύριο Νταφ ο οποίος προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση διότι ε, με, ε, από τον εκλογικό νόμο έχει περάσει πολύ καιρό και πρέπει να αναθεωρηθεί ο νόμος αυτός. Τώρα αναφερόμαστε στην πανευρωπαϊκή λίστα και η πολιτική μου ομάδα έχει υποβάλει μία τροπολογία επ' αυτού του θέματος γιατί ε, προσπαθούμε να προωθήσουμε με τον όρο αυτό που είχε ε, προ... Ε, παρουσιάσει για πρώτη φορά ο Ότο Φοχάσμπουργκ του οποίου τιμούμε τη μνήμη. Πιστεύω λοιπόν ότι 8 Μαΐου 1950 κάποιος θα είπε στο Σούμαν ή στον Αντενάουερ είναι πολύ νωρίς για να υπάρχει μία ε, γερμανογαλλική ΕΚΑΧ. Πάντοτε είναι πολύ νωρίς για όλους τους συντηρητικούς οι οποίοι δεν θέλουν θέλουν καμιά αλλαγή. Πάντοτε είναι πολύ νωρί. δεν είναι ποτέ ο κατάλληλο χρόνο. Για αυτού όμω που θέλουν να προχωρήσει η Ευρώπη, που έχουν όνειρα, μεγάλα όνειρα, και με πολλές προσωπικότητες πρέπει να έχει κανείς όνειρα υψηλά σαν τα βουνά κατά τρόπον ώστε να μπορούμε να κοιτούμε προς αυτά τα βουνά και σιγά σιγά να τα ανέβουμε. Χρειαζόμαστε έρευνα ιδεώδη ε, αγώνες γι' αυτό και το ΕΛΚ θέλει να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συνένεση σε αυτή τη γραμμή και αυτό θα κάνουμε. Όπως είπε και ο Πολ Βαλερή δεν σταματάει κανείς ποτέ εγκαταλείπουμε εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε θα επανέλθουμε κύριε Πρόεδρε Νίκο ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος και τώρα η κυρία Μπένοβα για ένα λεπτό Ευχαριστώ το βασικό στοιχείο ε, των διαπραγματεύσεων για την ε, αναθεώρηση της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήταν ότι δεν, ε, προβλέφθη, δεν προβλέφθηκε κανένας ενίος εκλογικός νόμος. και ε, στη, υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια στοιχεία μέσα στην έκθεση που μπορεί να φαίνονται προβληματικά, αλλά παρόλα αυτά ε, κάποια έχουν ήδη ρυθμιστεί και προτείνονται λύσεις. Έχουν διευρυνθεί οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1961 και μετά και χρειαζόμαστε νέα εσωτερική οργάνωση που να είναι στο ύψος των νέων αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Επίσης θα πρέπει να προσελκύουν οι εκλογές σε μεγαλύτερο βαθμό τους πολίτες. Ε, τώρα θα ακούσουμε την κυρία Γέτεν Μακή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου Άντριο Ντάφ. Δυστυχώς ε, διαπιστώνω παρόλα αυτά πως υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της έκθεσης που αδυνατόν να υποστηρίξω διότι αυτή η πρόταση για τους πρόσθετους 25 βουλευτές με τις διεθνικές λίστες είναι κάτι που είναι απαραίτητο να απορριφθεί. Είναι ήδη αρκετά μεγάλο το κοινοβούλιο. Έχουμε αρκετούς βουλευτές. Δεν είναι το πρόβλημα ο ρυθμός των βουλευτών. Το πρόβλημα είναι η αποτελεσματικότητα. Αν εργάζονται αποτελεσματικά. Πρόκειται για πραξικόπημα, κατά τη γνώμη μου, από πλευράς των μεγάλων κρατών μελών της Ένωσης. Ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών μας ε, συνίσταται στο να διατηρούμε στενές σχέσεις ε, με τους ανθρώπους που μας εκλέγουν. Και ο στόχος είναι αυτά τα, αυτοί οι 25 βουλευτές ε, ε, να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Δεν νομίζω όμως ότι είναι εφικτό. Ε, διωγώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς γίνεται δηλαδή να επισκέπτονται ε, και παραπάνω κάθε χώρα αυτοί οι 25 βουλευτές. Είναι ανέφικτο. Υπάρχουν άλλοι τρόποι ώστε να προωθήσουμε ε, ε, προεκλογικές εκστρατείες ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Δηλαδή μπορούμε ε, να βρούμε άλλους τρόπους δράσης. Τώρα ο κύριος Κοζούστνικ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ίνικο Μέντες, έναν φίλο και αγαπώ και τη χώρα του, αλλά παρόλα αυτά προθέλει να γίνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι πάρα πολύ έντονες σε αυτή τη φάση. Θυμίζω ε, την μειωμένη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ των πολιτών της Ευρώπης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θυμίζω επίσης ότι εμείς είμαστε το μοναδικό σώμα το οποίο εκλεγόμεθα άμεσα από τους πληθυσμούς της Ευρώπης και γι' αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργούμε συγχύσεις και περαιτέρω δυσκολίες. Εμείς προτείνουμε μέτρα, εμείς κάνουμε αλλαγές, αλλά οι πολίτες τι λένε, κανένας δεν ζητά την γνώμη των πολιτών. Οι ιδέες ακούγονται δεξιά και αριστερά, αλλά όλες αυτές οι ιδέες δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στους ευρωβουλευτές και αυτούς οι οποίοι τους εκλέγουν. Πολύ μεγαλύτερη απόσταση από ότι ανάμεσα στους εθνικούς βουλευτές και ε, τους εκλογές τους. Ευχαριστώ κύριε Νιούζικ. Χασί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι οι προσπάθειες που γίνονται για κάποιες μεταρρυθμίσεις είναι θετικές προσπάθειες. Συμφωνώ με τους περισσότερους από τους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στην έκθεση DAF. Παρ' όλα αυτά έχω κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την διεθνική αυτή εκλογική περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε μάλλον περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερο βάρος στις μεγάλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα κόμματα τα μεγάλα θα αποφασίζουν για το ποιοι θα είναι υποψήφοι και αυτό σημαίνει ότι μόνο εκπρόσωποι των μεγάλων κρατών μελών ουσιαστικά θα έχουν την δυνατότητα να εκλεγούν εφόσον τα ευρωπαϊκά κόμματα προτείνουν τους υποψηφίους αυτούς επαναλαμβάνω ότι θα προέρχονται από πολιτικά κόμματα των μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα αντικειμενικό σύστημα έτσι ώστε να ισορροπήσουμε το εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω να βρεθούν άλλες προτάσεις κύριε Ντάφ και άλλες λύσεις γιατί η πρότασή σας εδώ θα δημιουργήσει αύξηση του ευρωσκεπτικισμού. Κύριε Πρόεδρε, ε, στο πλαίσιο των ενεργειών μας του Κοινοβουλίου τίθεται το ερώτημα αν είμαστε επαρκώς νομιμοποιημένοι για τη δράση μας και ε, γι' αυτό ο κύριος Ντάφ με τη μακρά εργασία του και πήρα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και ε, πιστεύω το σημείο εκείνης του είναι σωστό ακόμη και αν όλες του οι προτάσεις δεν είναι υλοποίηση υλοποιήσιμες. Στην πολιτική μας ομάδα υπήρξαν συζητήσεις και προτάσεις οι οποίες αντικατοπτρίσουν το ενδιαφέρον και τις πείρες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ένα σημείο συμφωνούμε ότι ο χώρος για την απόφαση ε, δεν είναι μόνο το Κοινοβούλιο και γι' αυτό πιστεύω ότι αποδέχομαι την έκθεση αλλά θα πρέπει να κινηθούμε και προς το Συμβούλιο διότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δικιά τους φωνή και τα ευρωπαϊκά κόμματα πρέπει να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια αυτά. Ευχαριστώ τον κύριο Σόλτς και δίνω τώρα τον λόγο στον κύριο Ρώση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο παρά μόνο στρεφόμενοι στην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ομοσπονδιακού κράτους. Νομίζω ότι θα πρέπει να μην γίνει κάτι τέτοιο, να μην ελέγχεται η διαδικασία αυτή από μια ευρωπαϊκή αρχή. Είναι μια επιλογή η οποία δεν σέβεται τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ρίζες στην εκλογική τους περιφέρεια και θα προκαλέσει και υπερβολικό κόστος. Θα έχουμε άλλωστε στο τέλος δύο είδη ευρωβουλευτών θα έχουμε από τη μία κάποιους βουλευτές οι οποίοι θα πρέπει να γυρνάνε σε 27-28 κράτη-μέλη και δεν θα αντιμετωπίζονται φυσικά όπως οι άλλοι. Με τι ποσά θα μπορούν να καλύπτουν τα εδάφη τους. Ένα άλλο θέμα είναι η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διαγραφές από τον κατάλογο, η έλεγχη σε εκατομμύρια ε, ε, ψηφοφόρων. Αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Η δημιουργία ενός ενίου πολιτικού κόστους δεν θα πρέπει να φύξει την κυριαρχία των κρατών μελών. Εμείς πιστεύουμε στην Ευρώπη, την Ευρώπη όμως των λαών, μέσω των εκπροσώπων τους και όχι με ένα υπερκράτος αφεντικό και γραφειοκρατικό. Ευχαριστώ κύριε Ρώση. Τον λόγο έχει η κυρία Σίνκλερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρόταση αυτή δεν θα προσφέρει τίποτα στην ποιότητα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο τον πολίτη από τους πολιτικούς του. Ό,τι περιλαμβάνει η πρότασή σας είναι απαράδεκτη. Οι ποσοστώσεις για τα φύλλα είναι λάθος, οι θετικές διακρίσεις είναι λάθος. Εσείς έχετε κύριε Ντάφη υπολογίσει το κόστος της εφαρμογής των μέτρων. Όχι βέβαια η πρόταση αυτή είναι ανοιχτή σε σε Ένα βρετανικό κόμμα, το UKIP, λέει ελεύθερα και δημόσια ότι χρησιμοποιεί τα κοινοτικά χρήματα για την εθνική πολιτική του δράση. Η πρότασή σας είναι απαράδεκτη. Ο κύριος Καζίνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο λαός θεμελιώνει τη δημοκρατία. Λαός σημαίνει ταυτότητα, σημαίνει παράδοση, ενότητα, βούληση κοινή διακυβέρνησης. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ένα εκλογικό σύστημα είναι ένα μέσο το οποίο οικοδομεί έναν ευρωπαϊκό λαό, ένα ευρωπαϊκό δήμο. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Δήμος δεν είναι ακόμα εδώ μαζί μας και αυτό απεδείχθη στις τελευταίες ευρωεκλογές με την μείωση της συμμετοχής στις εκλογές. Και αυτό αποδεικνύεται επίσης και από το ότι οι εθνικές συζητήσεις γίνονται αυστηρά σε εθνικό επίπεδο και δεν αφορούν τα ευρωπαϊκά θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν μας υποχρεώνει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενιοποιήσουμε τις εκλογικές διαδικασίες. Δίνει την δυνατότητα. Η δυνατότητα αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν και δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αν θέλετε την προσπάθεια αυτή της μεταρρύθμισης της εκλογικής. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νταφ και σαν πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμικών Υποθέσεων η οποία έχει εγκρίνει το κείμενό της σχεδόν με ομοφωνία και ε, θα ε, μας στεναχωρήσει πολύ αν τεθεί εκ νέου σε συζήτηση. Νομίζω ότι παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο το οποίο να ε, μας δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη συνένεση. Υπάρχει ανάγκη ευρωπαϊκής αντίληψης των πραγμάτων όχι υποχρεωτικά από ένα ενιαίο εκλογικό χώρο, αλλά μέσω μεγαλύτερης εμπλοκής των λαών της Ευρώπης στην εκλογή των μελών και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή. Σας ευχαριστούμε κύριε Καζίνη. Τώρα η κυρία Ουλφσκουγκ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, υπάρχουν δύο προτάσεις μέσα στην έκθεση DAF που μπορούμε να ε, υποστηρίξουμε. Ε, νομίζω ότι πρέπει να σφιγμομετρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουμε τη θερμοκρασία για να καταλάβουμε αν θα αυξηθεί η προσέλευση στις εκλογικές αναμετρήσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέψουμε ένα από πιο συγκεκριμένο σύστημα για την εκλογή ε, των 25 αυτών βουλευτών. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η Επίτροπος ε, Δαμανάκη. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή την πρόταση ε, δεν έχουμε μακροπρόθεσμο ρεαλισμό. Είναι σαν να βλέπουμε τα πράγματα πάνω από ένα, μέσα από ένα ελικόπτερο. Νομίζω ότι είναι δουλειά των εθνικών κομμάτων να εξηγήσουν στους πολίτες ότι αυτά που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζουν θετικά ε, την καθημερινή τους ζωή. Δεν καταλαβαίνω πώς ένα έθνος, ένα κράτος μέλος μπορεί να σταθεί αντιμέτωπο ενώπιον των χρηματοπιστωτικών αγορών ή να υλοποιήσει μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αυτό μακροπρόθεσμα. Ας μην βλέπουμε βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο την έκθεση του κυρίου Ντάφαση. Είμαστε ρεαλιστέ. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό ο κύριο Δρινάλντι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, με την τροποποίηση αυτή επιβεβαιώνουμε δύο βασικές αρχές. Πρώτον, τον διευρωπαϊκό εκλογικό, την διευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό βήμα προς τον φεντεραλισμό και εδώ χαιρετίζουμε την επιμονή του εισηγητή. Αλλά ένας τέτοιος ε, εκλογικός κατάλογος ή καλύτερα μια τέτοια εκλογική περιφέρεια δεν θα πείσει τους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο. Απαιτούνται και άλλες παρεμβάσεις που θα μας φέρουν κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια δυναμική ανανέωση. Είχαμε καταθέσει μια τροπολογία, δεν έγινε δεκτή στην αρμόδια επιτροπή με γελίες δικαιολογίες. Ελπίζω ότι για την επόμενη ολομέλεια θα γίνουν και νέες προτάσεις σχετικά με τις περιφερειακές αλλαγές των εκλογικών περιφερειών έτσι ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση με την χώρα και τον τόπο προέλευσης. Από την άλλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκουαλτιέρη και την πολιτική του ομάδα έτσι ώστε να έχουμε ένα καθαρό κοινοβούλιο το οποίο να προβλέπει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα δεν έχουν δικαίωμα εκλογής. Για σοβαρά θα έλεγα προβλήματα όπως οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά, τρομοκρατία, φιλετική διάκριση λοιπά Τέτοιου είδους εγκλήματα δεν μπορεί να επιτρέπουν να είναι κανείς εδώ ευρωβουλευτής αν τα έχει διαπράξει. Μόνο αν είναι πρωτοπόρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκτήσει την αξιοπιστία που του αξίζει. Ευχαριστώ. Θα αρνηθώ την, ε, το μπλε δελτίο γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και έχουμε πάρα πολλού εγγεγραμμένου στον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Γκίρλινγκ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε θρίαμβε, ο κακός χρονισμός ως προς την ευαισθησία που δείχνουμε εμείς ε, απέναντι στους πολίτες ε, ενώ εκείνοι ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται πόσο κοστίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προτείνουμε ένα ακριβό νέο σύστημα για ε, μια νέα υπερδημοκρατία. Ένα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόστασης που ολοένα και μεγαλώνει ανάμεσα σε κάποιους βουλευτές και τους εκλογείς τους. Δείτε δείχνουν οι δημοσκοπήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι ευθύνη όλο ένα και περισσότερη υποστήριξη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και κυρίω για την ύπαρξη του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να αναστρέψουμε αυτή την τάση, θα πρέπει να βρούμε τρόπου να απηχούνται οι απόψει ε, των πολιτών ε, και άρα να ζητάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισηγείται ε, τι ενδεδειγμένε πρωτοβουλίε και να έχουμε μια προστιθέμενη αξία. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει ότι εμεί συντηρητικοί δεν έχουμε οράματα. Έχουμε. Θέλουμε μια προοδευτική Ευρώπη. Απλώ ε, τα δικά μα τα οράματα μα οδηγούν προ μια εντελώ διαφορετική κατεύθυνση, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι έγκυρα ε, και αν εσεί ακολουθήσετε τη ρότα που προτείνετε, θα μας ε, βοηθήσετε να επικρατήσουμε στο τέλος. Κυρία Σίνκλερ, έχετε ήδη μιλήσει εσείς και είναι μακρύτατο ο κατάλογο οπότε θα μιλήσουν αυτοί που δεν έχουν πάρει το λόγο. Ο Πάσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή της ε, και μετά μετεξελίσσεται δυναμικά και με κάποιο τρόπο εκπροσωπούνται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, οι πολίτες της Ένωσης ε, και με την εκλογική μεταρρύθμιση του 2014 όντως ή άλλως θα πρέπει να ασχοληθούμε και έχουμε πολύ συγκεκριμένε προτάσεις μέσα στην έκθεση του κυρίου Ντάφε και τις υποστηρίζω στην πλειοψηφία τους. Όμως ε, δεν είναι πολύ πρακτική η πρόταση αυτή για την θέσπιση 25 επιπροσθέτων εδρών στο Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με τον κύριο ε, Άντριου Ντάφ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε δύο διαφορετικά σώματα. Το σώμα των πολιτών που θα εδρεύει στις ε, Βρυξέλλες ε, με τις συνήθεις νομοθετικές και κοινοβουλευτικές εξουσίες του Κοινοβουλίου και ένα άλλο σώμα που θα έχει έναν αριθμό βουλευτών που θα υπολογίζεται βάσει ε, ενό ε, συντελεστή που ε, αυτή τη στιγμή μας οδηγεί σε τρει φορές 27 έδρες στο Στρασβούργο. Ε, φυσικά θα χρειάζεται κατάλληλο συντονισμό ανάμεσα στα δύο σώματα. διακόπτει η πρόταση, κυρία Ντότ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε πίτροπε. Αλλά δεν είναι περίεργο όσο ε, έχουμε τον ε, κύριο Κλέγκ του οποίου μειώνεται η συμμετοχή στην χώρα του να έχουμε τον κύριο Νταφ να προτείνει να αυξήσουμε τους ε, ευρωβουλευτές και αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι στιγμής οι εθνικοί βουλευτές δεν έχουν συνδέσει σωστά την Ευρωπαϊκή Ένωση με ε, τους ψηφοφόρους και εάν ζητούσε κανείς να υπάρξει πανευρωπαϊκή λίστα θα υπήρχε μία αρνητική απόφαση δεν, ε, διότι έτσι θα υπάρξουν όλο και μεγαλύτερες αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γι' αυτούς τους λόγους δεν υπάρχει ούτε διασύνδεση ούτε κατανόηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι ότου λοιπόν αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί κανείς να κυβερνά σαν αυτό σκοπό, και ε, ε, το να υπάρχουν επιπλέον 25 πανευρωπαϊκοί βουλευτές θα κοστίσουν περισσότερο και δεν θα έχουν καμία σχέση με την εκλογική τους βάση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ρασκόφσκι για δύο λεπτά. Αυτή είναι μία πρόταση φιλόδοξη την οποία καταρχήν πρέπει να στηρίξουμε. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα διότι ε, εφόσον υπάρξει μία διεθνική λίστα δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό άλλο. Υπάρχουν όμως λεπτομέρειες οι οποίες οδήγησαν στις ε, αντιρρήσεις. Είναι ένα πείραμα στην ε, φεντεραλιστική δημιουργία δημοκρατία για να δημιουργηθεί ένας ευρύτερος ευρωπαϊκός χώρος και πρέπει να στηριχθεί. Αν θέλουμε να είναι ορατά τα ευρωπαϊκά κόμματα, αν θέλουμε οι ψηφοφόροι να επιλέγουν βάση γνώσεων, εάν θέλετε δηλαδή ε, να αναλάβετε σωστά το ε, έργο σας και να το εκτελέσετε, πρέπει να ξέρετε τι κάνουν αυτά τα κόμματα. Θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές συζητήσεις συζητήσεις για ευρωπαϊκά θέματα και νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση αυτή. Εγώ είχα στηρίξει όταν ε, είπαμε να υπάρξει ε, πανευρωπαϊκή λίστα για να στηρίζουμε τους καλύτερους υποψηφίους και ε, εδώ ακούω στις μικρές χώρες ότι θα πρημοδοτηθούν τα μεγάλα κράτη δεν έχετε εμπιστοσύνη διότι αν οι Τσέχοι παραδείγματο χάρη έθεσαν, έθεταν τον Βάσλαβ Χάβελ πιστεύω ότι πολλοί θα τον ψήφισαν πολλοί οι οποίοι σκέφτονται σαν και εμένα αλλά αν βγάζαν τον Βάσλαβ Κλάους φαντάζομαι ότι ε, πολλοί συντηρητικοί θα τον ψήφιζαν και αυτόν δηλαδή υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτές τι ιδέε και ιδίω σε μια εποχή λιτότητος ε, δεν είναι το σωστό μήνυμα. Δεν ε, κάνει όμως απλώς πείσματα ο κύριος Νταφ. Είναι ε, κάτι το οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε βάσει πρωτοβουλίας. Έχουμε το δικαίωμα αυτό και ας το συζητήσουμε λίγο παραπάνω γιατί νομίζω ότι είναι μια αξιέπαινη πρόταση. Ωραία, ο κύριος Λένεν, Λάινεν ένα λεπτό. 30 χρόνια μετά από την πρώτη άμεση ε, ψηφοφορία χρειαζόμαστε μία ουσιαστική αλλαγή του συστήματος διότι δεν πρέπει ε, να μείνουμε ε, χωρίς να προχωρήσουμε και πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα δηλαδή να διατυπώσουμε το στρατηγικό εργαλείο της πανευρωπαϊκής λίστας. Η δημοκρατία είναι συζήτηση όπως έλεγε πάντοτε ο καθηγητής Αμερμάς και αυτό είναι το πρόβλημα. Η πολιτική τάξη έχει εθνικό διάλογο. Οι συζητήσεις περιορίζονται στον εθνικό χώρο και δεν έχουμε έναν μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο και θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να υποχρεώσουμε την πολιτική τάξη να κάτσει κάτω, να σκεφτεί, να συζητήσει, να επιχειρηματολογήσει ευρωπαϊκά και να δείξουν στους πολίτες ε, τι Ευρώπη μπορούν να επιλέξουν στις ευρωεκλογέ. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση του κυρίου Ντάφ είναι καλή και ε, είναι κάτι που το Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει ήδη δεν μπορούμε εμείς να οπισθοχωρούμε σε σχέση με τους προηγούμενους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Σμιτ τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Άντριο Νταφ, αρέσει πάρα πολύ η πρότασή σας γιατί θεωρώ ότι τροφοδοτεί τον προβληματισμό και είναι καλή για το μέλλον. Αλλά σχετικά σύντομα Μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση, αλλά τι σημαίνει αυτή η πανευρωπαϊκή λίστα, ότι θα τονιστεί η ευρωπαϊκή διάσταση της εκλογικής αναμέτρησης, ε, δηλαδή σαν να παίρνει σαν να παίρνουν βιταμίνες τα εθνικιστικά ε, κινήματα σε επίπεδο κράτους ε, μέλους. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να εξετάσουμε βαθύτερα το ζήτημα. Ε, εντάξει, να το ψηφίσουμε το χάβελε αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν καθόλου αυτοεπίθεση αυτοί που έρχονται από τις μικρές χώρες. Δεν το καταλαβαίνω. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες, συγγνώμη, έχουμε και Δανούς. Μικρή είναι η χώρα. Ο κύριος Κόξ έρχεται από την Ιρλανδία. Δεν ε, καταλαβαίνω. Έχουν την υποστήριξη από τα κόμματά τους. Μα ε, τονωθείτε, τονώστε την αυτοπεποίθησή σας. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές ε, και μπορούν να θεωρήσουν ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να ψηφίσουν δύο φορές ε, και να προωθήσουν τις πολιτικές που επιθυμούν σε επίπεδο ένωσης. Δεν χρειάζεται ε, να αλλάξει κάτι. Και θα ήθελα να πω προς την κυρία Ουλσκούγκ, ναι, να είμαστε ρεαλιστές, αλλά ορισμένε φορές ε, θα πρέπει λίγο να φύγουμε από την πεπατημένη, να είμαστε λίγο πιο θαραλέ. Είσαι πάρα πολύ συντηρητική Μαρίτα Ουλσκούγκ. Ευχαριστούμε κύριε Σμίτ. Ο κύριο Γιακολίνο τώρα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε το δικαίωμα στον Ευρωπαίο για τον Ευρωπαίο πολίτη θα πρέπει να κατοχυρώνεται και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε εκπρόσωποι των κρατών μελών και συγκεκριμένων εκλογικών περιφερειών είναι βασική θα έλεγα, είναι βασικό προνόμιο του κάθε Ευρωπαίου πολίτη να εκλέγει άμεσα τον εκπρόσωπό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε μορφή τροποποίησης της εκλογής των εκπροσώπων δεν θα πρέπει βέβαια σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι είναι κριτική ε, στις προτάσεις τις οποίες κάνει ο εισηγητής. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ναι μεν έχει σαν στόχο την καλύτερη και ενιαία εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Σώματος η δημιουργία μιας νέας εκλογικής περιφέρειας δημιουργεί θέματα σε σχέση με την εκλογή των Ευρωβουλευτών ως εκπροσώπων συγκεκριμένων περιοχών. Οι αρχές οι ευρωπαϊκές περνούν μέσα από την εφαρμογή της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της συνεργασίας ανάμεσα στην υπηρετική χώρα και τις νησιωτικές περιοχές και της αντιμετώπισης των άτακτων μερικές εποχές ε, μεταναστευτικών ροών. Ελπίζω λοιπόν κάποιες από τις τροποποιήσεις αυτές οι οποίες είναι συνεκτικές με την συναισθηματική αντίληψη μιας ενωμένης Ευρώπης να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο στόχος αυτός και με το καινούργιο αυτό, με την καινούργια αυτή πρόταση, την καινούργια εκλογική περιφέρεια. Ο Ευρωπαίος πολίτης θέλει να αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο σε αυτή την περίπτωση θα ταυτιστεί με τον εκπρόσωπό του και θα νιώσει εμπιστοσύνη. Και τότε μόνο θα έχουμε ένα οργανωτικό πρότυπο το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκλογέα. Ευχαριστώ. Ναι, θα προχωρήσουμε. Έχουμε μακρά, μακρά λίστα ομιλητών. Θα δώσω τον κύριο, στον κύριο Βαρσίδη τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πετύχουμε να ενδιαφερθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τα ευρωπαϊκά θέματα. Έγιναν διάφορες προσπάθειες στο παρελθόν για να βελτιωθεί το εκλογικό σύστημα και τώρα έχουμε τις εκλογές, τη, τη συζήτηση για τις εκλογές με ευρωπαϊκό κατάλογο, με ευρωπαϊκή λίστα. Ε, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μονομενοι υποψήφοι να υποβάλουν ε, τη δική τους υποψηφιότητα κλπ. Θα πρέπει επίσης να αντιδράσουμε σε αυτό που αναφέρθηκε που είναι μια επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωση και αποτρέπει την, ε, τον δημοκρατικό χαρακτήρα των εκλογών. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό εγώ δεν θα μιλήσω βουλγαρικά τη γλώσσα μου για να υπάρχει καλύτερη κατανόηση για την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ένα παράδειγμα ε, για τον εκθεμισμό. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ψηφίσουμε έναν, σε ένα ευρωπαϊκό κατάλογο. Οι λεπτομέρειες μετά πώς θα οργανωθεί αυτό, πώς θα πιστούν οι εκλογές ότι είναι σωστό, <clears throat> αν έχουμε φτάσει στο στη στιγμή, αν είναι σωστό να κάνουμε κάτι ή προσπαθούμε να μπλοκάρουμε. Η συγκεκριμένη αυτή ιδέα έρχεται σε μια σημαντική στιγμή. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να ε, εμβαθύνουμε, να δούμε κατά πόσον θα μπορέσουμε να αποφεύγουμε επανεθνικοποίηση. Ο Πολωνός Υπουργός χθες έβγαλε ένα λόγο πολύ πιστικό Και η έκθεση αυτή που έχουμε μπροστά μας ακριβώς αυτό λέει και είναι μια σημαντική πτυχή αυτού του οράματος. Κατά τη γνώμη μου, οι ευρωπαϊκές εκλογικέ λύσεις θα είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να είναι πιο ελκυστική η Ευρώπη. Αν απορρίψουμε αυτή την έκθεση θα είναι... Πρόεδρος Διακόπτη, παρακαλείτε να μιλάτε κάπως πιο αργά, κύριε Έλεγα λοιπόν ότι δεν θα καταλάβουν οι πολίτες της πατρίδας μας αν καταψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Ίσως αυτή η, έκθεση, η πρόταση δεν είναι ιδανική για πολλούς από μας, αλλά ας το συζητήσουμε, ας εξετάσουμε περαιτέρω την πρόταση αυτή. Ας έχουμε περισσότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών κομμάτων, ας έχουμε περισσότερη ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, ας από τους εθνικούς εγωισμούς. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα στην Ευρώπη και να της δώσουμε ε, μια εικόνα για τη δημιουργία αυτών των, <clears throat> των, ε, αυτής της εικόνας, αυτών των αναγκών. Θα πρέπει να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή προσώπηση και θα έχουμε υπέρ της έγκρισης έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Γρότε, ένα λεπτό, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Άντρου Ντάφ μας υπέβαλε μια οραματική και όπως είπε και ο ίδιος ριζοσπαστική πρόταση για την ε, μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος και μου ότι αυτό είναι πολύ καλό. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι διαφορετική. 18 συνάδελφοι περιμένουν να μπουν στο κοινοβούλιο και εμείς λέμε ότι θέλουμε να διευγρύνουμε το κοινοβούλιο με 25 συναδέλφους. Θα ήταν καλό αυτή η έκθεση, τη οποία τα περισσότερα σημεία υποστηρίζω, θα ήταν καλό να ξανασυζητηθεί ούτως ώστε να πετύχουμε ευρεία πλειοψηφία για την έκθεση αυτή η DAF στην τρίτη προσπάθεια. Γιατί χρειάζομαι, είμαστε ένα ενιαίο εκλογικό σύστημα και θα ήθελα πολλά από τα οράματα που παρουσίασε ο Άντρου Ντάφ κάποια στιγμή στο δεύτερο εξάμεινο του έτους να μπορούσαν να εγκριθούν και να εφαρμοστούν. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε ευρεία πλειοψηφία και όχι μικρή. Γιατί με μια μικρή πλειοψηφία δεν θα μας ακούσει κανένας. Ευχαριστώ κύριε Κρότε. Το λόγο έχει η κυρία του Χόνιστάιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι κατά την καμπάνια του Κοινοβουλίου είδαμε πόσο ο πολιτικός διάλογος επικεντρώνεται όχι μόνο στα εθνικά ζητήματα αλλά και σε τοπικά και όλοι συνειδητοποιήσαμε κατά την καθημερινή μας δραστηριότητα στις εκλογές μας περιφέρειας ότι δεν υφίσταται αίσθηση ε, του ότι όλοι ανήκουμε σε, στην ευρωπαϊκή οικογένεια και ότι ε, μας καίνε τα ευρωπαϊκά ζητήματα πόσο μάλλον ή πόσο λιγότερο απασχολείται ο κόσμος με τα ευρωπαϊκά κόμματα, κύριε Επίτροπε. Η συμμετοχή στις εκλογές, όχι μόνο για τις ευρωεκλογέ, μιλώ και για τις τοπικές, εθνικές εκλογές, ε, συνεχώς φθήνει, η αποχή αυξάνεται. Μεγάλο πρόβλημα. Και ποια είναι η λύση. Ε, όχι βέβαια να τους προτείνουμε λιγότεροι, αλλά περισσότερη Ευρώπη και θα πρέπει επομένω να αναβαθμίσουμε τον πολιτικό διάλογο για την Ευρώπη, τα πολιτικά συστήματα, να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες και αυτό είναι η πρόταση DAF. Εδώ μας κάνει μια αυθεντική συνεισφορά στην περισσότερη Ευρώπη, στη μεγαλύτερη Ευρώπη και τα είπε ο Πολωνός Υπουργός χθε και νομίζω ότι εκείνος εκπροσωπώντας το Συμβούλιο δηλαδή ένα θεσμικό όργανο διακυβερνητικό ότι είναι πιο κοινοτικό από ό,τι πολλές φορές το αυτό εδώ το κοινοβούλιο το οποίο είναι το κατεξοχήν εκπρόσωπών το κοινοτικό πνεύμα. Για να το σκεφτούμε αυτό, να το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε την πρόταση ΕΝΤΑΦ. Εγώ 100% συμφωνώ μαζί του. Η πρόεδρο, σα ευχαριστώ κυρία. Κυρία Οκονή, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα πρώτα Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο το οποίο επετέλεσε με την έκθεσή του και οφείλω να σας πω ότι και εγώ είμαι υπέρ ισχυρής Ευρώπης Ευρώπη που είναι προβεβλημένη Ευρώπη των λαών και είμαι φεντεραλίστρια. Θέλω επομένως να συστρατεύσουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε η Ευρώπη αυτή να γίνει πιο αποδοτική, πιο φιλόδοξη. Βεβαίω όμως και ξέρω ποιες είναι όλες αυτές οι δυσκολίες. Δυσκολίες του να εξηγήσω στους συμπολίτες μου, τους συμπατριώτες μου το ό,τι απασχολεί σήμερα τα θεσμικά όργανα μια που έχουν την αίσθηση οι συμπολίτες μου ότι έχουν αφαιθεί στο περιθώριο των εξελίξεων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε, δεν έχουμε την ελληνική κρίση, την κρίση του χρέους στην Ευρωζώνη, δεν έχουμε την πρόκληση για την βιομηχανία, την πρόκληση για τη βιομηχανία ε, τα 13 εκατομμύρια από αυτών των μη προνομιούχων οι οποίοι αναζητούν απελπισμένα κάποιες λύσεις ε, στις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Επομένω και εγώ θα πρέπει να κάτσω και να εξηγήσω στους κοντινούς μου αυτούς τους συμπολίτες το ότι πρώτα πρώτα ασχολούμαι με τα θεσμικά στο κοινοβούλιο. Επομένως και εγώ θέλω μια φεντεραλιστική Ευρώπη ε, και εγώ θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Ψοδέλτιο είναι ένα βήμα σημαντικό όμως σήμερα σήμερα να είπατε κύριε Ντεβίγκο να περιμένουμε αλλά πρέπει να εξηγήσω στον κόσμο ότι πρώτα πρώτα πρέπει να συζητήσουμε τα θεσμικά ενώ αυτοί ε, θεωρούν ότι έχουν αφαιθεί στο περιθώριο Βίλαντ Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε η συζήτηση εδώ αφορά ένα, μια οραματική ιδέα. Δυστυχώ έχουμε όμως τη συνθήκη τη Λισαβόνα όπου βλέπουμε ότι ξεπερνάει το κοινοβούλιο ότι το ρόλο του σαν ε, το δημιουργικό ε, σώμα της ε, Ένωσης. Δεν φτάνει στο ύψος αυτό των απαιτήσεων αυτή η έκθεση γιατί λέμε ότι θα υπάρχει πιο δίκαια κατανομή των εδρών. Σε τρία χρόνια από αρχή τη θα έχουμε το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα κριτήρια για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των μελών από τις μικρές χώρες. Αλλά αν βλέπουμε ότι ορισμένοι βουλευτές ε, προσωπούν 80.000 πολίτες και άλλοι βουλευτές εκπροσωπούν 800.000 και ότι εάν για κάθε πολίτη ο ένας ρίχνει την ψήφο του και κάνει πλικ, ο άλλος ρίχνει την ψήφο του και κάνει πλοκ, δεν είναι ισότητα δηλαδή αυτό το πράγμα. Στο παρελθόν μιλάγαμε για δημοκρατικό έλλειμμα γιατί δεν είχε τίποτα να λέει το κοινοβούλιο. Τώρα επιτρέπουμε ότι ε, μπορεί να επιτραπεί να λέμε ότι υπάρχει ε, δημοκρατικό έλλειμμα εάν δεν υπάρχει ζωστή αναλογία ανάμεσα στα μέλη του Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι που θα μας εγγυηθεί το μέλλον, άσχετα πώς θα είναι η εξέλιξη των αριθμών των πολιτών. Και έτσι δεν χρειάζεται πια να συζητάμε για ένα ε, δημοκρατικό έλλειμμα στο μέλλον. Συζητάτε, έχετε υποβάλει μια, ένα τύπο πολύ ε, περίπλοκο. Πώς θα μπορούν το 50% των ε, μαθητών να καταλάβουν ποια είναι η σύνθεση του Κοινοβουλίου. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye και δίνω το λόγο στον κύριο Νικολάζικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι όταν ξεχνάμε εδώ το θέμα του μεγίστου αριθμού των ε, εδρών ε, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένας ε, κίνδυνος γιατί αυτά είναι αριθμοί που είναι, στο, είναι εδρωμένα στην, στις συνθήκες. Εάν τώρα ανοίξουμε τις εκλογές, ίσως γνωστέ προσωπικότητε όπω τραγουδιστέ ποδοσφαιριστέ και άλλοι, ε, ε, γίνουν μέλη του Ευρωκοινοβουλίου χωρίς να εκπροσωπούν πραγματικά τη χώρα τους. Γιατί θα, από την άλλη μεριά θα έχουμε και γνωστές προσωπικότητες από μεγάλες χώρες μέλη που έτσι κι αλλιώς πολλά έχουν να πούνε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για τις μικρές ε, χώρες μέλη. Οι προσωπικότητες δηλαδή από τις μεγάλες χώρες μέλη είναι πιο γνωστές από εκείνες από τις ε, μικρές. Είναι γεγονός αυτό. Και τελειώνοντας, έχω να πω ότι θα πληγούν οι μικρές χώρες και γι' αυτό πιστεύω ότι το σημερινό σύστημα εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι νόμιμο και ε, αντιπροσωπεί πολύ την κατάσταση των ε, πολιτών. Η κυρία Τικάου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και τόσα χρόνια μετά την πρώτη εκλογή των Ευρωπαίων Βουλευτών βλέπουμε ότι δεν μας διέπουν ε, διευρωπαϊκές αξίες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Ε, οι ευρωβουλευτές που εκλέγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα, απόλυτη ισότητα, έτσι ώστε να εκπροσωπούνται και οι ε, ευρωβουλευτές σε αποδιακρατικούς καταλόγους, εκλογικούς καταλόγους. Θα πρέπει να θυμηθούμε το ρόλο των ευρωβουλευτών. Εκπροσωπούμε τις χώρες μας και τους και δεν θα πρέπει να προωθήσουμε ένα ελιτίστικο πλαίσιο τη στιγμή που δεν υπάρχει εκλογική βάση. Ολόκληρη η Ευρώπη θα είναι η εκλογική βάση και δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αιτιολογήσουμε μια τέτοια αλλαγή. Στόχος των Ευρωβουλευτών είναι να προωθήσουν την, ε, ε, την ελευθερία του εκφράζεσθε και ο καλύτερος τρόπος είναι με το σύστημα που έχουμε. Έχουμε ένα σαφή δεσμό με το εκλογικό σώμα και γι' αυτό αντιτάσσομαι σε μια τέτοια μεταρρύθμιση. Δεν νομίζω ότι είναι όριμη η καιρή για κάτι τέτοιο. Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε επιτέλους αυτή την πρόταση του συνάδελφου Ντάφ, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα βήμα προς την κατεύθυνση κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής. Όλοι εκλεγόμαστε σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό ε, αναρωτιέμαστε και μας ρωτάνε στις πατρίες μας τι είναι το σημαντικά εθνικό, όχι το ευρωπαϊκό. Εμείς έχουμε 25 ε, να έχουμε 25 βουλευτές που εκλέγονται ευρωπαϊκά συν τους άλλους είναι, έχει νομίζω νόημα. Και αυτό ως να μην γίνει βέβαια εις βάρος των μικρών. Εγώ προέρχομαι όμως από μια μικρή χώρα. Δεν έχω κανένα φόβο ότι θα χάσω, θα χάσω ψήφους. Δηλαδή θα υπάρχει ο καθένας ότι ε, έχει τη δυνατότητα να εκλέγεται ή σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο και εκλογικέ ε, περιφέρειε υπάρχουν έτσι και αλλιώ, Γιατί όχι για την Ευρώπη. Κύριε Βίλαντ, εσεί αναφερθήκατε σε αυτό το πολύπλοκο τύπο. Δεν υπάρχει όμω πάνω στην έκθεση. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε μια πρόοδο προ σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φιγκερέρο. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή βρίσκεται μακριά από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και διανύουμε μια στιγμή λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να, να εκλεγούν 25 επιπρόσθετοι ευρωβουλευτές. Και αυτό θα σταθεί υπέρ των μεγάλων κρατών, ξεχνώντας ότι έχουμε 27 κράτη-μέλη που μπορούν να εκλέξουν ευρωβουλευτές τους, ε, τους οποίους γνωρίζουν πολύ καλά και μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους άμεσα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να πλήξουμε τις μικρές και μεσαίες χώρες και το σύστημα άμεσης εκπροσώπησης, πραγματικής άμεσης εκπροσώπησης, μειώνοντας τη δημοκρατία και αυξάνοντας το ποσοστό αποχής στις εκλογές. Ο κύριος Στογιάννοφ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τι θα συμβεί όταν αποκτήσουμε αυτήν την ενιαία εκλογική περιφέρεια δεν είναι για καμία επιφύλαξη για τι καλέ προθέσει του κ. Νταφ. Όμω λένε ότι με τι καλέ προθέσει τρώνε το δρόμο προ την κόλαση. Επομένω, θα πρέπει να αποφύγουμε το να έχουμε ξαφνικά μια ολιγαρχία πολιτική που είναι επικυριαρχή. Θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να φροντίσουν να δουν πώ θα γίνει και δεν θα έχουμε κάποιο δυσυσόβια μέλη του Κοινοβουλίου μέσω αυτή τη λίστα. Ε, τι θα γίνει. Ξέρετε ότι όλο αυτό από τη μάτι θα κοστίσει 100 ευρώ παραπάνω για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τι θα γίνει επίση και με την εκπροσώπηση των εταιρικών μειονοτήτων στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνάδελφοι, αυτό που έχω να σα πω είναι ότι σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο έχουμε εδώ ένα δεδομένο αριθμό ε, γυναικών και ανδρών αυτών που αποφάσισαν να στείλουν οι εκλογεί, οι ψηφοφόροι. Τώρα, με την καινούργια ρύθμιση δεν θα ισχύσει το ίδιο. Κύριε Μέντε Δεδίου, έχετε, έχετε το λόγο. Ο κύριος Κουτσίνσκι που δεν είναι πλέον στην αίθουσα είπε κάποιου χαρακτηρισμού Είπε ότι ε, ε, ε, είμαι θεροβάμων καλύτερα όμω παρά να ζω στο παρελθόν σαν κι αυτόν. Ναι, μα είπατε ότι εδώ πέρα συζητάμε, η κυρία από τη Γαλλία, συζητάμε θεσμικά και όχι πραγματικά. Ναι, όμω ένα Γάλλο, Ζαν Μονέ, είπε ότι τα θεσμικά όργανα χαράσουν την πολιτική. Κυρία μου, σήμερα μόλι, πριν αυτή τη συζήτηση, κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Αυτή η άλλη συζήτηση αφορούσε την, το, το, το, τη διανομή τροφίμων στου φτωχού. Δηλαδή, βλέπετε ότι όλα γίνονται, όλα γίνονται με, με, με κάποιο έφτακτο τρόπο. Επομένω, και αυτή η ιστορία λέτε ότι η λίστα είναι κατά των μικρών χρόνων. Εμεί όμω λόγω του Σαντέρ, τότε είχαμε το Γιούγκερ, ε, όλους αυτούς, αυτοί από πού έρχονται οι πρόεδροι της Κομισιόν. Ε, όχι πια. Προσοχή, προσοχή, δεν θέλω μέσα κατά του Λουξεμβούργου, λέει η πρόεδρος. Αλλιώς θα, θα, θα, θα έχετε πελάτε. Κύριε Σοκοντή, κύριε Πρόεδρε, η συνιστόσα γαλλική στο ΕΡΚ σε ευρία πλειοψηφία είναι κατά τη ενιαίας λίστα του ενιαίου ε, ψηφοδελτίου βουλά πολιτική, οικονομική κλπ. Διότι σήμερα έχουμε όλα τα θεσμικά όργανα ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α προσέξουμε επομένω να μην ε, μπλέξουμε την, την, την επιτάχυνση ε, την αποτελεσματικότητα με την βιασύνη γιατί σήμερα συζητούμε για κάποιο είδους εκλογές ε, το 2014 το πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω στα χέρια μας έχουμε κάθε μέσο τόσο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την ευρωπαϊκή ιδέα οπότε θα πρέπει να μην βιάζεται το ε, κοινοβούλιο θα πρέπει να γίνονται τα εθνικά κοινοβούλια, Σέγγεν, ε, Κυβερνήσει, διακυβέρνηση. Δεν έχουν μπορέσει να συσπηρώσουν τα βρετή πλειοψηφία. Όμω ε, τώρα προσπαθούμε να ε, φτιάξουμε κάποια κατασκευάσματα αντικοινωτικά. Α είμαστε, είμαστε πιο υπομονετικοί. Δεν υπάρχει σήμερα η κατάλληλη συγκυρία για τον φεντρεαλισμό που μια μέρα θα το πετύχουμε. Επομένω, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρί. Ε, να προχωρούμε με γρήγορα βήματα, αλλά όχι βιαστικά. Ευχαριστώ. Κέλλη. αντιτίθεμαι σε αυτή τη σύσταση σε σχέση με τους επιπρόσθετους ευρωβουλευτές παρόλο που θαυμάζω τον κύριο Νταφ. Το γεγονός ότι θα είχαμε 25 επιπρόσθετους ευρωβουλευτές που θα τους εκλέγουν όλοι αλλά δεν θα είναι υπόλογοι σε κανέναν δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια τέτοια κατάσταση ιδιαίτερα σε καιρούς ύφτεσης όπου για παράδειγμα στη χώρα μου έχουμε μειώσει τους βουλευτές, μιλάμε για κατάργηση του δεύτερου σώματος, μείωση των βουλευτών μας και τώρα μιλάμε για 25 επιπρόσθετους ευρωβουλευτές. Αυτό είναι άκερο και άσκοπο. Θα πρέπει να λογοδοτούμε στους πολίτες ακόμα περισσότερο λεπτό. Η, λέξη δημοκρατία σημαίνει ε, κυβέρνηση των λαών. Λαών ω σύνολο. Δεν σημαίνει κυβέρνηση από έναν αυθαίρετο αριθμό ανθρώπων, διότι δεν μπορούν να ασκήσουν τη δημοκρατία. Διότι δεν υπάρχει αμεσότητα μία διευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια δεν είναι κάτι το οποίο να τύχει αναγνώρισης. Ίσως να φτάσουμε σε μια τέτοια ταυτότητα, αλλά η ταυτότητα αποτελεί πρόκριμα και δεν είναι απότοκη μιας εκλογικής διαδικασίας. Μόνο τα ευρωπαϊκά ε, μόνο τα, η ευρωπαϊκή αυτή οντότητα προβάλλεται έναντι των κρατικών. Ε, τότε κάποια στιγμή θα μας πείτε ότι τον, το ίμιση των ευρωβουλευτών ή το εν τρίτον θα πρέπει να εκλέγεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να δράσουμε υπέρ των ευρωκρατών. Η κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο για να γνωμοδοτήσει ως προς την ε, ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση πράγματι μια και μίλησα επί μακρόν, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με εκείνους που θεώρησαν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών για ευρωπαϊκά ε, ζητήματα και να τους ενθαρρύνουμε να ψηφίζουν στις εκλογές. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να βελτιώσει αυτό το πλαίσιο, το περιβάλλον, δηλαδή των επόμενων ευρωεκλογών. Αναφερόμενοι στην εκλογική μεταρρύθμιση, όπου το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας, θα ήθελα να πω ότι αναμένουμε την σύνοψη της συζήτησης με βάση την έκθεση DAF και θα επέμβουμε στη συνέχεια. Κύριε Ντάφ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ε, εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς ε, εκείνους που παρευρέθησαν στη συζήτηση και παρέμειναν για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα πολιτικής εμβέλειας ως προς το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ιδιαίτερα επίκαιρο. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η λίστα που προτείνεται, η πανευρωπαϊκή, θα λογοδοτεί, θα λογοδοτεί απόλυτα στο κοινό, στην κοινή γνώμη. Ιδιαίτερα στην εκλογική εκείνη βάση η οποία έχει κουραστεί ιδιαίτερα από, τις, από την εθνική πολιτική, από τις εθνικές πολιτικές. Νομίζω ότι είναι κάτι το ευκταίο και η πρόταση αυτή θα πρέπει να αναπεμφθεί στην Επιτροπή για, για να την σκεφτούμε καλύτερα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, διευρύνουμε αυτή την εντολή μέσα στα πλαίσια της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου και της συζήτησης με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα και για να διευρύνουμε το πλαίσιο των υποστηρικτών, των ευρωπαϊστών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Νταφ και σας ευχαριστώ όλους για αυτή την μακρά και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η ψηφοφορία δεν θα γίνει σήμερα γιατί θα αναπαιμφθεί το θέμα στην Επιτροπή. Τώρα θα συζητήσουμε την έκθεση